των κειμένων θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Πριν περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση, η κυρία Μπατσελή, ε, Κράμερ, ε, Κοχμερίν και τα λοιπά για τους ειδικού Ολυμπιακούς ε, Αγώνες συνέλεξε υπογραφές των μισών και πλέον βουλευτών και πάνω από, σύμφωνα με το άρθρο 116, θα δημοσιευθεί και θα διαβιβαστεί στους ε, αποδέκτες. Σύμφωνα με την ημερησία δίδυξη, ακολουθούν τώρα δηλώσει Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την κατάσταση δημοκρατία τη Μολδαβία. Αλλά ο κύριο Γότσον κάτι θέλει να πει, γιατί έχουμε εξέχοντε Μολδαβού εδώ παρόντε σήμερα. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στην παρουσία στο